Good afternoon, ladies and gentlemen. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καθίστε παρακαλώ. Μπορούμε να αρχίσουμε. Είμαστε αρκετοί, αρκετά μέλη της Επιτροπής Περιφερειακών Υποθέσεων και φαντάζομαι ότι σύντομα θα έρθουν και άλλοι στην αίθουσα και άλλοι συνάδελφοι. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχετε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης για τη σημερινή συνεδρίαση, σωστά. Έχω κάποιες παρατηρήσεις. Οι μας, η συγγητρία μας μάλλον για το Omnibus, η κυρία Κρέλ, θα μας ενημερώσει στα διάφορα για ό,τι έχει γίνει στον τριμερή διάλογο. Αυτό θα γίνει αύριο στο τέλος της συνεδρίασης. Οπότε στα διάφορα έχουμε ήδη αυτό το σημείο για αύριο. Αν δεν υπάρχουν άλλες προτάσεις, σχόλια, τότε εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Συνεχίζουμε με την έγκριση των πρακτικών τη συνεδρίασή μας στις 7 Σεπτεμβρίου. Το σχέδιο πρακτικών διατίθεται online ως ήθιστε. Αν δεν έχετε αντιρρήσεις κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης, τότε θεωρούνται εγκεκριμένα. Αν έχετε αντιρρήσεις, σχόλια θα μου το πείτε. Επόμενο θέμα. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Έχω κάποιες ανακοινώσεις. Και αρχίζω με το ότι σήμερα υπήρξε μια ανοιχτή συνεδρίαση για την εβδομάδα Περιφέρειες και Πόλεις. Και εγώ είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την Επιτροπή μας μαζί και με τον κύριο Λάμπερτς που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών και η κυρία Κορίνα Κρέτσου, επίτροπος ήταν παρούσα. Σήμερα άρχισε η 7η αναθεώρηση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με κάποια μηνύματα για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Επίσης, Συμμαχία της Συνοχής είναι μια νέα πρωτοβουλία που αρχίζει προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι, οι μαρχές, οι τοπικές, οι περιφερειακές, οι πολιτικοί, όλοι μαζί να συμμετέχουν σε μία συμμαχία για την εξέλιξη της πολιτικής συνοχής στο μέλλον. Αυτά έγιναν σήμερα και γι' αυτό και αρχίζουμε αργότερα τη συνεδρίασή μας από τη συνήθως. Η επόμενη πληροφορία που έχω να σας δώσω έχει να κάνει με το εργαστήριο που οργανώνει ΣΤΟΑ Πρόκειται για την Κοινοβουλευτική Υπηρεσία για την Επιστήμη και την Τεχνολογία. Ποιε είναι οι επιλογέ και πώ γίνεται η αξιολόγηση. Οργανώνουν λοιπόν ένα εργαστήριο για τι νέε τεχνολογίε και την περιφερειακή πολιτική προ την επόμενη πολιτική συνοχή. Αυτό θα γίνει τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου. 2.30 έω 6.30 το απόγευμα. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην αίθουσα Α5Ε2. Ζητάω από τη Γραμματεία να στείλει όλες αυτές τις πληροφορίες στα μέλη της Επιτροπής μας, ώστε αν θέλουν να παρευρεθούν στο εργαστήριο αυτό. Βασίζεται το εργαστήριο αυτό σε προτάσεις που έστειλε η ίδια η Επιτροπή μας στην ΣΤΟΑ το 2015, όπου ετοιμάσαμε κάποιες γνωμοδοτήσεις, κάποιες, κάποια σχόλια, τα οποία στείλαμε και στη ΣΤΟΑ. Και να τώρα έχουμε το εργαστήριο που θα ασχοληθεί με αυτά. Τώρα ο κύριος Φανίστερο και η κυρία Κρέλ θα προεδρεύσουν ε, τις δύο συνεδρίες του εργαστηρίου αυτό με τον κύριο Βαλκαφέρε Σίσο που και τον αντιπρόεδρο, ο αντιπρόεδρος της ε, ΣΤΟΑ θα αναλάβει την ε, κήρυξη των εργασιών, ο κύριος Πυρίνσκι. Σαν μέλος της ΣΤΟΑ επίσης θα κλείσει το εργαστήριο αυτό. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη της Επιτροπής μας όσο, όσοι θέλετε να πάτε. Θα σας ενημερώσει η Γραμματεία με περισσότερες λεπτομέρειες και ελπίζω ότι η συμμετοχή της Επιτροπής μας θα είναι ευρεία. Γιατί πρόκειται για θέματα το που έχουν να κάνουν με το δικό μας έργο. Το δεύτερο, η δεύτερη πληροφορία που έχω να σας δώσω έχει να κάνει με την συνεδρίαση της ε, Επιτροπής Προέδρων των Επιτροπών 26 Σεπτεμβρίου και 3 Οκτωβρίου. Μετά από την ομιλία του κύριου Γιούνκερ για την κατάσταση πραγμάτων στην Ένωση και την επιστολή του, οι πρόεδροι επιτροπών συνεδρίασαν με τους ομολόγους τους από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συνεδρίαση αυτή οργανώθηκε σε ομάδες ανάλογα με τα θέματα πολιτικής και τις ιδέες που θέλαμε να συζητήσουμε σε σχέση με το πρόγραμμα της Επιτροπής για το 2018, το οποίο έγκριση προβλέπεται για την 24η Οκτωβρίου. Οι ομάδες αυτές λοιπόν συνεδρίασαν 26 Σεπτεμβρίου με 3 Οκτωβρίου και στο τέλος είχαμε και μια ολομέλεια στις 3 Οκτωβρίου, όπου προέδρευαν από κοινού η κυρία Βίλκστρομ από πλευράς της Επιτροπής Προέδρων Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον κύριο Τίμερμαν από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στι 26 Σεπτεμβρίου, τώρα, εγώ συμπροείδρευσα στην ομάδα Επενδύσει, Απασχόληση και Ανάπτυξη. Μαζί με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις διάφορες επιτροπές, την οικονομική, απασχόληση περιβάλλοντος, σύμκο και πολιτισμού. Ο κύριος Κατάινεν συμπρόδευε μαζί μου από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον συνούδευαν οι Επίτροποι Τομπρόφσκης, Τίσεν, Βιενκόφσκα, ναβράσις, Κρέτου, Φεστάγερ και Μόιντας. Στις 3 Οκτωβρίου συμμετείχα στην ε, ομάδα που συνεδρίασε με θέμα ε, μελλοντική χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με τους πρόεδρους της Επιτροπής Προπολογισμών, τον κύριο Αρτουής και της ε, Κόντ, Ντεβε, Απασχόληση, Ήτρε, Μεταφορές, Γεωργία, Πολιτισμός και Λίμπε. Όπως καταλαβαίνετε, όλες αυτές οι ομάδες συζήτησαν για ένα σωρό θέματα πολιτικής. Για μας σημασία είχε, είχαν οι επενδύσεις στην Ευρώπη υπέρ της πολιτικής συνοχής που έχουν πολύ καλή απόδοση αποτελούν μια προστιθέμενη αξία, ιδιαίτερα όταν συνδέονται και με τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Υπογράμμισε επίσης ότι οι επενδύσεις σε προγράμματα υποδομών είναι ζωτικής σημασίας γιατί βοηθούν το ανθρώπινο δυναμικό, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την ε, διοικητική ικανότητα. Χρηματοδότηση λοιπόν, χρηματοδοτικά μέσα είναι συμπληρωματικά μέσα και δεν αποκλίνουν το ένα το άλλο. Και είναι αυτά τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν παρετέρω. Δύο είναι τα συμπεράσματα. Πρώτον, ότι οι προτάσεις για την νέα γενιά προγραμμάτων πρέπει να υποβληθούν ε, την άνοιξη πριν το καλοκαίρι, ώστε να μπορέσει να τα επεξεργαστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν από τις εκλογές του 2019. Και το δεύτερο συμπέρασμα ήταν ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις συνεργασίες μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στατικών Επενδύσεων, για παράδειγμα, και των επενδύσεων για τον ε, ορίζοντα 2020 και όχι μόνο. Αυτά λοιπόν είναι τα κύρια μηνύματα που έχω να σας μεταφέρω από αυτήν τη συνάντηση. Πρέπει επίσης να σας πω ότι πολλοί συνάδελφοι και εγώ μεταξύ άλλων, εκφράσαμε τις ανησυχίες μας για το γεγονός ότι το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο άργησε να ετοιμαστεί εν ώψη της άνοιξης καλοκαιριού 2020. Εμείς θα έχουμε στη διάθεσή μας λιγότερο από 10 μήνες για να δουλέψουμε πάνω σε αυτές τις προτάσεις πριν τις εκλογές, έτσι, του 2019. Συνεπώς, το χρονοδιάγραμμα αρχίζει και γίνεται πολύ σημαντικό στοιχείο. Ακούσαμε τις αντιδράσεις της Επιτροπής, αλλά αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι ο Αντιπρόεδρος και ο Επίτροπος Έτιγκερ ακολουθούν αυστηρά τον χάρτη πορείας που περιλαμβάνεται στην επιστολή του Πρόεδρου Γιούνκερ προς τον Πρόεδρο Ταγιάννη. Οπότε το δημοσιονομικό πλαίσιο εμείς πρέπει να το περιμένουμε από ό,τι φαίνεται το Μάιο του 2018. Έτσι έχουν τα πράγματα. Αυτά λοιπόν τα συμπεράσματα της συνάντησης αυτής των διαφόρων ομάδων και της Ολομέλειας όπου συμμετείχαν οι πρόεδροι Κοινοβουλευτικών Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με επιτρόπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το τελευταίο που έχω να σας πω είναι για αποστολή στη Ρουμανία. Όπως ξέρετε, την πρόσφατη πράσινη εβδομάδα η Επιτροπή μας έστειλε μια αντιπροσωπεία στο Κλούσου Απόκα που είναι η δεύτερη μεγάλη πόλη της Ρουμανίας. Εκεί ακολούθησαν ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα συναντήσεων και επισκέψεων, που μεταξύ άλλων επισκέφθηκαν και ένα ορυχείο, δεν βλέπω τον κύριο Τσέλερ εδώ, ο οποίος προείδρευε της αντιπροσωπείας αυτής, αποστολής της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να μας ενημερώσει περισσότερο για την αποστολή αυτή, αλλά κάποια άλλη στιγμή θα το κάνουμε όταν θα είναι εδώ. Δεν τον βλέπω. Αυτές ήταν οι ανακοινώσεις που είχα να σας κάνω για σήμερα. Και μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να περάσουμε σε Επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση επί της απόφασης 189 του 2014 του Συμβουλίου με την οποία επιτρέπεται στη Γαλλία να εφαρμόσει μειωμένο συντελεστή για ορισμένου έμεσους φόρους στο παραδοσιακό ρούμι που παράγεται στη Γουαδελούπη, τη Γαλλική Γουιάννα, τη Μαρτινίκα και την Ίσο Ρεϊνιόν και με την οποία καταργείται η απόφαση 2007-659. Η συγγήτρια για το θέμα αυτό είμαι εγώ ίδια. Και πρέπει να σας πω να σας πω το παραδοσιακό ρούμε της Γαλλίας από τις απότερες ε, περιοχές από το 1923 υπόκειται σε ε, ειδικούς φόρους κατανάλωσης και ειδικές διευθετήσεις για τη γαλλική αγορά ε, την υπηρετική. Όμως η αγορά του ρουμιού παγκοσμίω αυξάνεται και οι ποσότητες του επιλέξιμου προϊόντος για ειδική φορολογική μεταχείριση περιοδικά προσαρμόζονται για να αντιμετωπιστεί η μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα του τομέα αυτού που έχει να κάνει με το ρούμι από ζαχαροκάλαμο για τι απότερε περιοχέ τη Γαλλία. Το 2016 η παραγωγή ρουμιού τη Γαλλία από τις εξόχου από απόκεντρες περιοχές ξεπέρασε την επιλέξιμη ποσόστοση για ειδική φορολογική μεταχείριση κατά 1 πέμπτο. Εάν η ποσόστοση του 2016 αλλάξει αναδρομικά δεν θα υπάρχει πρόβλημα, Ιδάλω η παραγωγή θα υποστούν οικονομική ζημιά. Το Σεπτέμβριο του 2016 οι γαλλικέ αρχέ ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μία ένα σχέδιο τεχνικής προσαρμογής για την πιο πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου αυξάνοντας την ετήσια ποσόστοση από 120.000 σε 144.000 εκτόλιτρα καθαρού αλκοολούχου ποτού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσάρμοσε την πρότασή της στις 9 Ιουνίου 2017 Είμαι η εισηγήτρια για το θέμα αυτό. Όταν οι συντονιστέ συζήτησαν την πρόταση, η άποψή του ήταν ότι δεν ήταν αμφιλεγόμενο και ότι μπορούσε να εγκριθεί χωρίς τροπολογίες βάσει της απλουστευμένης διαδικασία. Βάσει του άρθρου 50, εδάφιο 1. Τώρα, μετά, ε, βάσει με αυτής της διαδικασίας, θα δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές για τον τοσχέ αυτό. Εάν έχουν παρατηρήσεις να κάνουν ή παρατηρήσεις ή για τη διαδικασία ή για τον τοσχέ το ίδιο, για το θέμα. Να ξεκινήσω με τον κύριο Πόγκα, ο οποίος μιλά εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω, Νομίζω να εφαρμόσουμε την απλουστευμένη διαδικασία και ώστε δυνατόν ταχύτερα να εγκρίνουμε το σχετικό κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανσχούρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, να χαιρετήσω την απόφαση του Συμβουλίου αλλά και την προσπάθεια του Επιτρόπου, του κυρίου Πιέρ Μοσκοβισή, ο οποίος μας, μας επιτρέπει με αυτήν την προσαρμογή να ε, ανανεώσουμε την αφοσίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υποστήριξή της προς την παραγωγή νοηματοδών από ζαχαροκάλαμο ε, στις εξόχως απόκεντρες ε, περιοχές της Γαλλίας. Ξέρετε ότι βάσει το άρθρο 359 τη Συνθήκη Λειτουργία για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για το θέμα αυτό, ε, είναι υπεύθυνο το Συμβούλιο. Και υπ' αυτήν την έννοια, σωστά το είπατε, Πρόεδρε, πρόκειται για μια τεχνική προσαρμογή τη απόφαση του Συμβουλίου που εξοσοδοτεί το παραδοσιακό Ρωμαίο από τι εξόχω απόκριτε περιοχέ τη Γαλλία να υπόκειται σε ειδικέ φορολογικέ διθετήσει. Είναι μια τεχνική προσαρμογή πολύ σημαντική γιατί αφορά την αύξηση των ποσοστώσεων που θα περάσουν από 120.000 εκτόλιτα σε 144.000 με αναδρομική ισχύ. Αυτή η προσαρμογή είναι μια αποτελεσματική απόκριση, θεωρώ, γιατί ο, η δυναμική ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς του ρουμνιού ε, ωφελεί περισσότερο του παραγωγούς των τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν διαφορετικές κοινωνικές και περιβαλλοντικέ ε, προδιαγραφέ. Πολλέ φορέ πολύ απομακρυσμένες από τα πρότυπα που αναγκάζονται να ε, ακολουθήσουν οι Ευρωπαίοι παραγωγοί. Υπ' αυτήν την έννοια, η ετήσια ανανέωση και προσαρμογή της ποσόστοσης για το ρούμι από τις εξόχους απόκεντρες περιοχές της Γαλλίας, Ντομπτόμ, είναι πραγματικά μια ανάσα για την οικονομία των εξόχω απόκεντρων περιοχών τη Γαλλία. Σε αυτέ 40.000 θέσει εργασία, εμέσω και αμέσω. ε, και ένα μεγάλο μέρος των γεωργικών εξαγωγών σχετίζονται με αυτόν ακριβώς τον τομέα. Ε, θα συμφωνήσω λοιπόν με τον κύριο Πόγκα. Ελπίζω να εγκριθεί πολύ γρήγορα το κείμενο αυτό για να τεθεί σε ισχύ ήδη από την αρχή της επόμενης χρονιάς. Ευχαριστούμε. Αυτή ήταν και η πρόθεση των συντονιστών όταν προτείναμε την απλουστευμένη διαδικασία. Ο κύριος Φλακ από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η απόφαση αυτού του Συμβουλίου είναι πολύ σημαντικό θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω για τους ε, συναδέλφους. Τουλάχιστον τρεις από τους σκιώδεις εισηγητές εκπροσωπούν Γάλλους ε, υπηκόους που ζουν εκτός της υπηρετικής Γαλλίας. Οι συντηρητικοί και μετρηθμιστέ συμφωνούν ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη τι ανάγκε των εξοχώ αποκεντρών περιοχών τη Γαλλία. Ωστόσο, να επιστήσω την προσοχή σα στο γεγονό ότι έχουμε κάποιε ίσονο σημασία επιφυλάξει. Πρώτον, οι σύμβουλοι μου είναι ιδιαίτερα απογοητευμένοι που για την ώρα δεν είχαμε καθόλου δείγματα ή κάποια κοινοποίηση από κάποια επίσκεψη για να συγκεντρώσει στοιχεία επιτόπου. Ε, αυτό είναι κάτι που μας λείπει. Επίσης, κατά δεύτερον, πιστεύουμε ότι όλα τα μέτρα προστασίας τη αγορά, πρέπει να είναι κατάλληλα για το σκοπό που επιδιώκουν, Ένα σκόπιμα. Το, η παραγωγή του ρουμιού είναι ένας βιομηχανικό κλάδος ανταγωνιστικός διεθνώς και θα πρέπει η Γαλλία ε, ειδικά ε, να αυξήσει βάσει αυτή τη απόφαση κατά 24.000 ε, εκτόλιτρα καθαρού ενοπνεύματος την ποσόστοσή τη. Ελπίζουμε, ε, καθότι αυτό είναι σκόπιμο, να μην υπάρξει καμία στρέβλωση τη αγορά κατά τα άλλα και προβλήματα αλλού. Η, το αίτημα της Επιτροπής, η παραδοσιακή ποσόστοση του 2016, ε, η απόφαση για αυτή την προσαρμογή της παραδοσιακής ποσόστοσης, να γίνει με τον κατάλληλο τρόπο και το άρθρο 349 της συνθήκης προβλέπει ίση μεταχείριση για όλε τι και τι εννέα εξοχώ απόκεντρε περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Να είμαι σαφή δηλαδή, οι συντηρητικοί και οι μεταρρυθμιστέ δεν έχουν ένσταση ε, να στηρίξουν συγκεκριμένε περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Απλώ θεωρούμε ότι το άρθρο 449 είναι άδικο, διότι καλύπτει μόνον εννέα συγκεκριμένε εξόχω απόκεντρε περιοχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι δεν είναι πάντοτε δίκαιη η μεταχείριση των περιοχών αυτών και η πυροτική Ευρώπη κάποιες φορές μπορεί να ε, την χάνει άλλης μεταχείρισης λόγω κλιματικών, τοπογραφικών συνθήκων. Και επίσης πρέπει να δούμε και τι διατάξεις περιέχουν ε, κανονισμοί για τα διευθυντικά ταμεία ε, και μπορεί να χρησιμοποιηθούν εδώ. Πρόεδρε, πάντοτε ήμουν υπέρ των προτάσεων για τη μείωση των φόρων στα αλκοολούχα ποτά. Ευχαριστούμε. Ήταν πολύ σαφής και πολύ ανοιχτή η τοποθέτησή σα. Δεν βλέπω τον κύριο Μαρεζέ, ο οποίο είναι ο άλλο σκιώδη εισηγητή. Κάποιος άλλος που θέλει να πάρει το λόγο εκ μέρου του. Ωραία. Ο κύριο Ροπέ. Όχι. Δεν είναι εδώ. Ο κύριος Μάτο δεν είναι ούτε εκείνος εδώ. Κάποιος άλλος Θέλετε το λόγο για τη διαδικασία ή το θέμα. Ωραία. πρόταση δεν είναι αμφιλεγόμενη. Στηρίζεται την παραγωγή ρομιού. Θα προτείνω λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει με την απλουστευμένη διαδικασία όντω, χωρί τροπολογίε, βάσει του άρθρου 351 και να εγκρίνει την πρόταση σε αυτή την συνάντηση. Έχει κάποιος αντίρρηση. Όχι. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, θα συμπεριληφθεί στον κατάλογο των ψηφοφοριών σήμερα η πρόταση. Α, δεν χρειάζεται καν. Εγκρίθηκε. Ωραία. Εγκρίθηκε βάσει της αποστευμένης διαδικασίας και θα ελπίσουμε να προχωρήσουν τα πράγματα όσο ταχύτερα γίνεται. Ευχαριστούμε τους σκιώδεις εισηγητές και πάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η ετήσια έκθεση για τις οικονομικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Καθήλυνα αρμόδια είναι η Επιτροπή Προπολογισμών. Η δική μας εισηγήτρια είναι η κυρία Μάλετιτς. Η ε, κυρία ε, Μάλετη θα μας παρουσιάσει σήμερα το σχέδιο γνωμοδότησής της. και προτείνω προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 12 ε, η ώρα την 3η 17 Οκτωβρίου βάσει και του χρονοδιαγράμματος της Καθήλυνα Αρμοδίας Επιτροπής. Κυρία Μάλετη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Με μεγάλη μου χαρά ανέλαβα την σύνταξη αυτής της γνωμοδότησης για αυτές τις πολύ σημαντικές ε, δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που ε, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την υποστήριξη της ε, εφαρμογής της πολιτικής συνοχής και επίσης όσον αφορά την ενίσχυση των ικανοτήτων για την προετοιμασία των έργων, την, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και την προετοιμασία των εθνικών ε, συγχρηματοδοτικών προγραμμάτων. Η ΕΤΕΠ λοιπόν διαδραματίζει πολλούς σημαντικούς ρόλους, ε, επιτελεί πολλούς ε, στόχους και έχει μια πλειάδα δραστηριοτήτων που αναλαμβάνει από την συμβουλευτική υποστήριξη, την ανάλυση με επικεφαλής τον Τζέρμι και τον, και τον Τζέσικα, ε, την ε, δανειοδότηση, ε, άμεσα δάνεια, παγκόσμια δάνεια, ενδιάμεσα δάνεια, δάνεια πλαίσια, συγχρηματοδοτικά μέσα και κτλ. καθώς και τις δραστηριότητες ενίσχυσης ικανοτήτων μέσω της πρωτοβουλίας Jasmine. Για να μπορεί να παρακολουθεί και να εκτιμά την συμβολή της ΕΤΕΠ στην πολιτική συνεχής, χρειαζόμαστε εμείς ως Επιτροπή ε, ειδικά κεφάλαια. Διότι χωρίς αυτά δεν μπορούμε να παρακολουθούμε ούτε να αξιολογούμε όλες αυτές τις διαδραστηριότητες που υλοποιούνται σε διάφορα κράτη-μέλη. Και το κεφάλαιο αυτό, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να αφιερώνεται στις δραστηριότητες ΕΤΕΠ που έχουν ως στόχο την ε, υποστήριξη της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής, αλλά θα πρέπει αυτό να γίνεται από τα κράτη-μέλη ε, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για την χρήση των ε, δανείων που χορηγεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επίσης δεν υπάρχουν δεδομένα όσον αφορά τα, ε, έργα που δανειοδοτούνται μεταξύ άλλων και από τα ε, ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Χωρίς αυτή την πληροφορία δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε την συμβολή της ΕΤΕΠ στην ε, εφαρμογή της πολιτικής συνοχής. Επίσης, αυτό που πρέπει να υπογραμμίσουμε ιδίω είναι το γεγονός ότι η ΕΤΕΠ πρέπει να συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων που έχουν τεθεί σε, ευρωπαϊκή, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην οικονομική εδαφική ε, συνοχή. Ωστόσο, βάσει της γεωγραφικής ανάλυσης της δανειοδότησης προς τα κράτη-μέλη, προς τα οποία δηλαδή ε, ε, ε κατευθύνονται τα δάνεια υπάρχουν μόνο 5 κράτη-μέλη στα οποία κατευθύνονται το 54,12% όλων των ε, δανείων που χορηγήθηκαν το 2015. Σχεδόν το μισά δηλαδή, πάνω από το μισά δηλαδή, ε, πήγε σε 5 ε, κράτη. Ξέρουμε ότι δεν υπάρχει γεωγραφική ποσόστοση για τη δανειοδότηση από την ΕΤΕΠ. Ωστόσο η συγκέντρωση αυτή σε 5 μόλις κράτη-μέλη καταδεικνύει ότι δεν μπορεί κανείς να πει ότι οι δραστηριότητες της ε, ΕΤΕΠ υποστηρίζουν την ε, οικονομική, πολιτική και εδαφική συνοχή είναι ένα στοιχείο που πρέπει να βελτιωθεί και να αλλάξει ως προς την ε, δραστηριότητα της ΕΤΕΠ. Επίσης, πάνω από το 50% των εγκριθέντων δανείων έχουν επενδυθεί στις, μεταφορές, μεταφορές, στην ε, ενέργεια και στις εσωτερικές πλωτές οδούς. Κάτι που δείχνει και μια θεματική συγκέντρωση. Αν δούμε όμως την ε, γεωγραφική κατανομή, από το συνολικό ποσό που ε, κατευθύνεται στη βιομηχανία, το 82% κατευθύνεται τελικά σε 5 κράτη-μέλη. Και στην ενέργεια το 72% επίσης πηγαίνει πάλι σε αυτά τα 5 κράτη-μέλη. Ενώ από το ποσό που κατευθύνεται στις μεταφορές, το 58% και πάλι ε, πηγαίνει σε αυτά τα κράτη-μέλη. Υπάρχει λοιπόν μια γεωγραφική κατανομή που ε, χαρακτηρίζεται από ανισομετρία. Κατευθύνεται κατά κύριο λόγο σε αυτά τα πέντε κράτη-μέλη. Πρέπει επίσης να δούμε πώς θα βελτιώσουμε το ρόλο της ΕΤΕΠ όσον αφορά τις νεοφυείς επιχειρήσεις, ε, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, τη γενική ε, επιχειρηματικότητα και θα πρέπει οπωσδήποτε η διαδικασία να απλουστευτεί και να αυξηθεί ο αριθμός των χορηγούμενων δανείων. Επίσης πρέπει να επιδιώξουμε να βελτιώσουμε και να αυξήσουμε τα έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΤΕΠ σε αγροτικές, σε εξόχως απόκεντρες, σε ε, ε, ε περιοχές ε, χαμηλής ανάπτυξης. Αυτά θα πρέπει όλα να αποτελέσουν προτεραιότητες όσον αφορά την χρηματοδότηση των έργων από την ΕΤΕΠ. Επίσης, ο ρόλος της ΕΤΕΠ στην πολιτική συνοχής αυξάνεται τα τελευταία χρόνια, ιδίως λόγω της αυξημένης χρήσης των χρηματοδοτικών μέσων. Η χρήση βεβαίως ε, αυτών των χρηματοδοτικών μέσων είναι ακόμη πολύ χαμηλή ε, και τα κράτη-μέλη επικαλούνται την ε, συνθετότητα και την περιπλοκότητα των διαδικασιών για το χαμηλό αυτό επίπεδο. Βεβαίω γνωρίζουμε ότι η ΕΤΕΠ δεν είναι εκείνη που καθορίζει τις διαδικασίε. μπορεί όμως να ε, συντάξει μια έκθεση όσον αφορά τα αρνητικά και τα θετικά στοιχεία της διαδικασίας αυτής και με, από τεχνική άποψης να υποστηρίξει την χρήση και την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Και κάτι τελευταίο που σχετίζεται με τα ευρήματα της μελέτης για την αναθεώρηση του ρόλου της ΕΤΕΠ όσον αφορά την Ευρωπαϊκή ε, Πολιτική συνοχή που συνέταξε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων όπου και διαπιστώνεται η έλλειψη δεδομένων όσον αφορά τον ρόλο της ΕΤΕΠ σε κάθε ε, κύκλο εφαρμογής των, πολιτικών, ε, των, των προγραμμάτων πολιτικής συνοχής. Ε, στην επιλογή, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, σε όλους αυτούς τους διάφορους κύκλους της εφαρμογής των προγραμμάτων δεν είναι σαφής ο ρόλος της ΕΤΕΠ. Και αυτό ε, αποδεικνύει σε όλους ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει πιο εντατική και συχνή επικοινωνία με την ΕΤΕΠ, ενώ και η ίδια η ΕΤΕΠ θα πρέπει να ε, βελτιώσει το δικό του σύστημα υποβολής εκθέσεων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στον τομέα της ε, πολιτικής συνοχής. Ε, βεβαίως σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διαφάνεια αλλά και την ορατότητα των δραστηριοτήτων της. Ευχαριστούμε κυρία Μάλετιτς. Ας δώσουμε τώρα το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Η κυρία Τόμασιτς θα εκπροσωπήσει τον κύριο Πορέλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την πολιτική συνοχή, είναι ένας ρόλος ο οποίος από 2000 και μετά έχει ενισχυθεί πολύ, ιδιαίτερα μετά την εισαγωγή ειδικών μέσων όπως είναι το Τζέσικα, το Τζάσπερ και το Τζάσμεν. Ήδη από το 2007 στο 2013 διαπιστώσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει συμμετάσχει πάρα πολύ στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Υπάρχει συγχρηματοδότηση για διάφορα προγράμματα συνοχής με δάνεια, κάτι πολύ σημαντικό ως κλίμακα και στηρίζονται με αυτόν τον τρόπο όλα τα προγράμματα πολιτικής συνοχής σε μεγάλο βαθμό. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συνεισφέρει λοιπόν στους στόχους της πολιτικής συνοχής και ε, με υψηλό επίπεδο προστιθέμενης αξίας. Οι χώρες μέλη θεωρούν ότι οι δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι αποτελεσματικέ όσον αφορά την απορρόφηση, για παράδειγμα, αλλά και τα αποτελέσματα. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση και αναλυτική στήριξη και τεχνογνωσία είναι στοιχεία κλειδί μέσω των οποίων συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα στην υλοποίηση της πολιτικής συνοχής. Όμως υπάρχουν περίπλοκοι κανόνες υψηλό ο κόστος της διαχείρισης είναι οι κύριε προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αυτό πάντως που με ικανοποιεί είναι ότι υπάρχει ε, τεχνική αρρωγή για όλα τα χρηματοδοτικά μέσα. Είναι κάτι που συνεισφέρει στην οικοδόμηση ικανοτήτων και βοηθάει τους ενδιάμεσους όλες τις χώρες μέλη. Ρόλος της τράπεζας αυτής ενισχύεται στην ε, πολιτική συνοχής. Έτσι υπάρχουν και διαφορετικές δραστηριότητες που δεν γίνονται πάντα κατανοητές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρχει λογοδοσία βέβαια ε, για τα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και έλεγχος της συνεισφοράς της τράπεζας αυτής ε, προς την πολιτική συνοχή που πολλές φορές η συνεισφορά αυτή είναι κατακαιρματισμένη και η ανάλυση της. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βέτεμπορκ. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σίγουρα έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει μια που συμπληρώνει τα οικονομικά μέσα τη χρηματοδότηση, αλλά και τους στόχους της πολιτικής συνοχής. Τα χρηματοδοτικά μέσα που έχουν αναπτυχθεί, έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και η αποτελεσματικότητα ε, των μέσων αυτών έχει αμφισβητηθεί πολλές φορές και από την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου. Ε, υπάρχει ελάχιστη ανάλυση για το πόσο συνεισφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με τα νέα αυτά χρηματοδοτικά μέσα. Όσον αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης, το στηρίζουμε γενικά. Ευχαριστούμε και την εισηγήτρια και επιφυλασσόμεθα να συντάξουμε τροπολογίες προκειμένου να ενισχύσουμε τη σημασία που έχουν τα χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για την πολιτική συνοχή, αλλά όχι μόνο και για την έρευνα και για την ανάπτυξη και πρέπει να αναπτύξουμε μηχανισμούς που να βοηθούν και στα πλαίσια του Ιντερεκ. Γιατί θα αποκτήσουν όλο και μεγαλύτερη σημασία την επόμενη περίοδο. Προσβλέπω λοιπόν σε συνεργασία με την Ιβάνα που είναι η συγγήτρια. Γιατί είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό και για την πολιτική συνοχή μετά το 2020. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Σκελετ δεν είναι εδώ, κύριος Μάτο δεν είναι εδώ. Άλλος κανείς που θέλει το λόγο για αυτό το θέμα. Όχι. Έχουμε εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως εδώ. Ο κύριος Σότο. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Όχι. Όχι. Όχι, ευχαριστούμε. Καλώς. Εντάξει, ευχαριστεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι εντάξει με τη γνωμοδότηση αυτή. Οπότε θέλω να σας υπενθυμίσω προθεσμία για υποβολή τροπολογιών είναι στις 12 το μεσημέρι στις 17 Οκτωβρίου, 3η 17 Οκτωβρίου. Φροντίστε λοιπόν. Α, συγγνώμη όμως, μια στιγμή. Έχουμε εκπρόσωπο εδώ τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Μήπω εσείς θέλετε το λόγο, ο κύριο Ντεμάντ. Ευχαριστώ, <clears throat> κύριε Πρόεδρε. Ναι. Και ευχαριστώ την εισηγήτρια, την κυρία Μάλεντιτς και όλους τους σκιώδεις εισηγητές που σχολίασαν και αναφέρθηκαν στην γνωμοδότηση αυτή. Εσείς στήξατε πολλά σημαντικά ζητήματα για την τράπεζά μας και θα αναφερθώ σε μερικά μόνο από αυτά. Αλλά σίγουρα ε, κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της τελικής γνωμοδότησης θα επανέλθουμε. Πρώτα απ' όλα, τι ακριβώς κάνουμε για να στηρίξουμε την πολιτική συνοχής. Όπως υπόθηκε, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την τράπεζά μας και ο ρόλος μας είναι να στηρίξουμε την υλοποίηση της ευρωπαϊκής πολιτικής και άρα να στηρίξουμε την πολιτική συνοχή που αποτελεί μία από τις προτεραιότητές μας. Τα τελευταία δέκα χρόνια πρέπει να ξέρετε 200 δισεκατομμύρια χρηματοδοτούμε περίπου για προγράμματα υπέρ της πολιτικής συνοχής. Από το 2000... Το 2016 μάλλον έχουμε δώσει λίγο λιγότερο από το 30% των δανείων που δίνουμε για την πολιτική συνοχή. Άρα αποτελεί προτεραιότητα για την τράπεζά μας και θα εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα και στο μέλλον η πολιτική συνοχή για μας. Το άλλο που θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι δεν προσφέρουμε μόνο χρηματοδότηση, αλλά βοηθούμε και τις περιφέρειες με συμβουλές και τεχνική αρρωγή. Άρα δεν βοηθούμε μόνο με χρηματοδότηση, βοηθούμε και την προώθηση του προγραμματισμού στις διάφορες περιφέρειες και πόλεις για να ετοιμάσουν σωστά τα προγράμματά τους και άρα η υλοποίησή τους να είναι επιτυχής. Όπως αναφέρθηκε ήδη, Βοηθούμε επίσης τις περιφέρειες να απορροφήσουν τα διορθωτικά ταμεία. Έχουμε κάποια συγκεκριμένα ε, εργαλεία Συγχρηματοδοτούμε προγράμματα διαρθρωτικών ε, ταμείων σε επίπεδο περιφερειών. Έτσι στηρίζουμε και την υλοποίηση προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα ένα χρηματοδοτικό μέσο δεν αποτελεί πανάκια, όμως Έχουμε υπόψη μας ότι μπορεί να υπάρξει ακόμα βελτίωση για να διευκολυνθεί η χρήση των χρηματοδοτικών αυτών μέσων. Γνωρίζετε όλοι ότι στην επόμενη περίοδο πολιτές δημοσιονομικές προοπτικές θα υπάρχει μείωση του προϋπολογισμού και για την στήριξη της περιφερειακής πολιτικής, οπότε τα χρηματοδοτικά μέσα θα αποκτήσουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Γι' αυτό τώρα που αναφέρατε προηγουμένως για τη γεωγραφική ισορροπία. Η Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων βελτιώνει το εύρος στο οποίο δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς όμως δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ζήτηση εκεί που δεν υπάρχει ζήτηση. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να δούμε πού υπάρχουν προγράμματα και να τα αξιολογήσουμε ανάλογα με το πόσο καλά είναι. Είναι ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων επίσης να βοηθήσει να συμβουλεύσει σε διάφορες πόλεις και περιφέρειες εκείνους οι οποίοι εκπονούν προγράμματα για να μπορέσουν να υποφεληθούν όσο γίνεται περισσότερο από χρηματοδότηση. Κάτι άλλο που είναι σημαντικό βέβαια είναι η στόχοι της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όταν μιλάμε για πολιτική συνοχή, φυσικά και στόχος της τράπεζάς μας είναι να βοηθήσει τις πόλεις και τις περιφέρειες ακριβώς για να ανταποκριθούμε στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το τελευταίο το οποίο αναφέρθηκε ήταν κάτι για τις κοινωνικές συνέπειες, τον κοινωνικό αντίκτυπο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για την ομάδα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, δηλαδή και του Ταμείου και της Τράπεζας. Προσπαθούμε να διοχετεύσουμε ε, κεφάλαια κινδύνου για τις startups, για παράδειγμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Μαλέτη, Θέλετε να απαντήσετε. Σας ευχαριστώ όλους. Συμφωνώ απόλυτα ότι όντως στην έκθεση θα πρέπει να υπάρχουν παραπάνω στοιχεία. Αλλά υπάρχει, βλέπετε, ένας περιορισμός ε, στην έκταση του κειμένου, γι' αυτό δεν μπορούσα να τα καλύψω όλα στο σχέδιο αυτό γνωμοδότησης. Αλλά με τις τροπολογίες μπορούμε μαζί να συμπληρώσουμε τη γνωμοδότηση αυτή. Μπορούμε να προσθέσουμε κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αστική πολιτική, το ίντερεγκ, τις διάφορες ε, μακροπεριφερειακές στρατηγικές κλπ. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που υπογράμμισε τη σημασία που έχει το να καταφέρουμε να κάνουμε κάπως διαφορετική τη γεωγραφική κατανομή και πολύ σωστά λέτε ότι έχετε ως ρόλο να βοηθήσετε αυτούς που ε, σχεδιάζουν τα προγράμματα και θα έπρεπε να δούμε πώς θα μπορέσουμε να δουλέψουμε περισσότερο πάνω σε αυτό με χώρες οι οποίες δεν συμμετέχουν και τόσο πολύ στη δανειοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ξέρετε, προθεσμία για τροπολογίες, το είπαμε. Και τώρα συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη και περνάμε στη συζήτηση ε, της γνωμοδότησης, συντάκτρια γνωμοδότησης είναι η κυρία Σμόλκοβα, η οποία είχε κάποια προβλήματα με τις πτήσεις της, οπότε ο κύριος Πίκοβα θα παρουσιάσει τη γνωμοδότηση αυτή. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρου τη εισηγητρία, τη κυρία Μόλκοβα, θέλω να διαβάσω τι σημειώσει τη για το θέμα. Να εκφράσω την εκτίμησή μου για την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι προτάσει τη για νομοθετική δράση στον τομέα τη ε, καθαρή ενέργεια για όλου και τη σχετική πρωτοβουλία. Η μετάβαση προ την καθαρή ενέργεια και τον τομέα αυτό ε, προσδοκάται να ε, να απτυχθεί στο μέλλον και πρέπει να επενδύσουμε σε αυτόν. Οι επενδύσει στην καθαρή ενέργεια είναι ένα θέμα που αφορά τον καθένα πολίτη και την κάθε μια από του πολίτε ξεχωριστά. Θεωρώ ότι είναι ύψη τη σημασία γιατί στόχο είναι να βελτιώσει την ποιότητα τη διαβίωσή μα η επιτυχία της ανάπτυξης καινοτομιών στον τομέα της ενεργείας αφορούν όχι μόνο τις εταιρείες, εταιρείες ενέργειας, ε, κατασκευαστικές ή ε, πληροφορικής, αλλά και αυτούς που παράγουν εξοπλισμό, τους παρόχους, ε, τις μεταφορές, όλους τους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και ιδρύματα και τις δημοτικές αρχές καθώς και τη δημόσια δίκηση. Να τονίσω ευθύ εξ αρχής ότι είναι τεράστιο το φάσμα των θεμάτων που καλύπτονται από τις καινοτομίες της καθαρής ενέργειας. Η γνώμη μου να σε οκτώ σημεία, τα οποία βρίσκω σημαντικά για τη δουλειά της Επιτροπής μας για την Περιφερειακή Ανάπτυξη. Ωστόσο, για να μην ξεχνάμε και το ιστορικό αυτής της τομέας, θα έλεγα να σταθούμε σε τέσσερις τομεί που αφορούν το περίπλοκο θέμα των κοινοτομιών στην καθαρή ενέργεια. Πρώτα απ' όλα, χρηματοδότηση. Είναι ένα τομέα όπου τα διευθυντικά ταμεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα επενδυτικά ταμεία μπορούν να συμβάλλουν. Ζητούμε αύξηση στον προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη τη πολιτική ενέργεια, ώστε σε συνεργασία με την ΕΤΕΠ και τη, τα ιδιωτικά κεφάλαια να συμβάλλουμε ώστε να υπάρξει ακόμη περισσότερη και επιταχυμένη καινοτομία στον τομέα τη ενέργεια. Δύο, η επιστήμη και η έρευνα. Ιδίω ό,τι αφορά τι στρατηγικέ καινοτομίε, οι ευφυεί πόλει και οι λύσει του παρουσιάζουν ανάγκη για πραγματικό συντονισμό των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Με προγράμματα εθνικά των κρατών μελών, εκεί που υπάρχουν επικαλύψει και επαναλήψει, να χρησιμοποιούνται με δραστικότερο τρόπο όλα τα μέσα για την καινοτομία τη καθαρή ενέργεια που μπορεί ήδη να χρησιμοποιούνται. Η συνεννόηση και ανταλλαγή των πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών περιφερειών και περιοχών λείπει σε αυτό το τομέα η ανάπτυξη της έννοιας της εφιούς εξειδίκευσης στα πλαίσια της συνοχής πολιτικής της πολιτικής συνοχής 2014-2020 είναι ο σωστός δρόμος. Όμως πρέπει να υπάρξουν περισσότερες διαπεριφερειακές εταιρικές σχέσεις μεταξύ των οποίων εταιρικές σχέσεις στον τομέα της ε, πολιτικής ενέργειας. Τρία. Οι πολίτες και η καθοριστική τους ε, θέση στην διαδικασία κοινοτομίας της ε, πολιτικής καθαρής ενέργειας. Όχι μόνο ως καταναλωτών της ενέργειας αλλά και ως παραγωγών της. Πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες ότι οι διαδικασίες καινοτομία θα φέρουν ε, εξοικονομήσεις και πλεονεκτήματα καθώς και προστασία του περιβάλλοντος. Υπό αυτή την έννοια οι πολίτες μπορούν να παίξουν ένα καθοριστικό ρόλο στα πλαίσια της ε, ατζέντα για τα αστικά κέντρα διότι ε, έτσι θα καταλάβουν καλύτερα τις συγκεκριμένες ευκαιρίες από τις επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας καθώς και το πώς μπορούν να επηρεάσουν οι ίδιοι. Ε, αυτό έχει ως σημαντικότερη επιτυχή την προσέγγιση bottom-up. Τέσσερα. Ο συντονισμός και η απλούστευση. Όλα τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ορίζοντας 2020, το ε, στρατηγικό ταμείο και τα διαθωτικά ταμεία, καθώς και το ε, Διευθυντικά Ταμείο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη επιτρέπουν περισσότερη απλούστευση και καλύτερο συντονισμό στη δικαιούχη που εφαρμόζουν συγκεκριμένα έργα και προγράμματα να έχουν άμεση πρόσβαση στις πηγές χρηματοδότησης. Τέλος, η κυρία Σμόλκοβα θέλει να ευχαριστήσει τη γραμματεία της Ρέντζε για τη στήριξή της και ανυπομονή για τις τροπολογίες σας και την περαιτέρω συνεργασία μας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την στήριξη και τα καλά λόγια της κυρίας Σμόλκοβα. Τώρα να δώσω το λόγο στους Σκιώδης. Κύριε Ντέλη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να επενέσω την εισηγήτρια για την πολύ καλή της δουλειά και εκ μέρου του ΕΛΚ να κάνω μια-δυο παρατηρήσεις. Κατά πρώτον, η καθαρή ενέργεια και η μείωση των εκπομπών είναι μια σημαντικότατη αρμοδιότητα όλων μας, ένα σημαντικότατο καθήκον. Και το να περικόψουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι ένα καθήκον παγκόσμιο, όχι μόνο δικό μας. Μάλιστα το ποσοστό της Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου ε, στο 11% αυτή τη στιγμή σε σχέση με το σύνολο. Πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας. Και όταν θα διατυπώσουμε για τις παρατηρήσεις μας επί της έκθεσης το είχαμε υπόψη. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι τα κέντρα καινοτομίας και η κατανομή τους συνήθως συγκεντρώνονται στα περισσότερα αναπτυγμένα, στα πιο προηγμένα μέρη της Ευρώπης, όπου ούτως ή άλλως υπάρχουν ερευνητικά κέντρα, που μειώνουν ούτως ή άλλως τις εκπομπές δραστικά και ήδη συμμετέχουν στην ενεργειακή μετάβαση. Εμείς ως Επιτροπή Ρέτζι πρέπει να αναφέρουμε σαφώς ότι χρειάζεται και άλλε πιο απομακρυσμένε περιοχές και λιγότερο αναπτυγμένε περιοχές να συμμετάσχουν σε όλη αυτή την προσπάθεια, ώστε να καλύψουν την απόσταση που τις χωρίζει από τους πρώτους σε αυτόν τον τομέα. Τρίτη παρατήρηση, λίγο πιο χειροπιαστή. Σημεριζόμαστε την προσέγγιση της εισηγήτριας ό,τι αφορά τη σημασία των κονδυλίων για την ενεργειακή μετάβαση στην Ευρώπη αλλά θα πρέπει τα διαφορετικά ταμεία να διατηρήσουν ανέπαφο το ρόλο τους για την πολιτική συνοχή. Και τέταρτη παρατήρηση, με συγχωρείτε το πέμπτη, είναι ότι και πάλι συμμεριζόμαστε πλήρως ε, την ε, έμφαση που δίνει η συγκήτρια στην προσέγγιση bottom-up, από κάτω προς τα πάνω. Ε, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία, ξεκάθαρη σημασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ζωτικό ρόλο να διαδραματίσουν σε ό,τι αφορά την καινοτομία στην ενέργεια και το να βγουν οι καινοτόμε λύσεις από τα εργαστήρια στους δρόμους για να χρησιμοποιηθούν. Αυτά από εμάς θα φροντίσουμε να αποστείλουμε τις τροπολογίες μας σχετικά. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιον από τους υπόλοιπους σκιώδεις. Α, ο κύριος Βανότεμπορκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να κάνω κάποιες παρατηρήσεις εκ μέρους της δικής μας εισηγήτριας, της κυρίας Νικολάη. Πρώτα απ' όλα η καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και η επιτάχυνση τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλή κατανάλωση άνθρακα είναι μια από τι βασικέ προκλήσει τη Ευρώπη. Από αυτή την έννοια, όλου και όδε πιστεύουμε ότι έρευνα και ανάπτυξη μέσω του ιδιωτικού τομέα είναι μια λύση ιδίω μέσω των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έτσι θα στηρίξουμε την καθαρή ενέργεια και θα βελτιώσουμε καθώ και θα επιτρέψουμε την δημιουργία θέσεων απασχόληση και την οικονομία τη Ευρώπη. Πρέπει να προσαρμοστούμε στι ανάγκε των πολιτών. Αυτή τη στιγμή, βάσει των επίσημων δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα από του πρωταγωνιστέ και του μεγαλύτερου χρηματοδότε τη έρευνα και ανάπτυξη στην καθαρή ενέργεια και τη σχετική καινοτομία. Υπάρχει όμω περιθώριο βελτίωση. Η εισηγήτριά μα συμφωνεί απολύτω με την εισηγήτρια επί τη ιδέα ότι είναι ποικιλόμορφη και πολύπλοκη χρηματοδότηση και τα εργαλεία τη ώστε σε αυτή τη φάση. Ορίζοντα 2020, διευθυντικά ταμεία, Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Αναβιώσιμη ε, Ανάπτυξη και το καθεξής. Επίσης, υπογραμμίζει την ανάγκη απλούστευσης πρόσβασης στη χρηματοδότηση για τις τοπικές αρχές, τις δημοτικές αρχές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ένα άλλο θέμα που επισημαίνει είναι ότι το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 μπορεί να διδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην έρευνα, την ανάπτυξη και να δώσει όθηση στην κοινοτομία, ενθαρρύνοντα και επιταχύνοντα τη μετάβαση σε αγαθά και προϊόντα, σε προϊόντα και υπηρεσίε που επιτρέπουν τη δημιουργία ανάπτυξη νέων θέσεων οικονομική ανάπτυξη και ε, πλούτο θα πρέπει να ακολουθήσουμε την προσέγγιση της ε, στοχευμένης ε, επιδότησης των ορυκτών καυσίμων μόνο σε ειδικέ περιπτώσεις και να επιδιώξουμε το στόχο μας με μια ενέργεια, με οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα και ενεργειακά ευφύ, με τη συνεργασία όλων εταιριών, μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, ε, ενδιαφερομένων, καταναλωτών. Όλες αυτές, όλες αυτές οι προσπάθειες συντονισμού πρέπει να υποστηριχθούν για να καταλήξουμε στη σωστή λύση. Πρέπει να εντοπίσουμε και να καταπολεμήσουμε την γραφειοκρατία, το διοικητικό άκτος, αλλά και τις τρευλώσεις στην αγορά, τις άδικες πρακτικές στην αγορά τις αθέμητες μάλλον πρακτικές. Διότι δεν συνάδουν με το αναδυόμενο πρόσωπο των καινοτόμων λύσεων. Επίση, για την απαλλαγή από τον άνθρακα πρέπει να ανακαινιστούν πολλά ευρωπαϊκά κτίρια και γενικότερα να σεβαστούμε τι πραγματικέ προδιαγραφέ. Με την προστασία των ειδικών προστατευόμενων περιοχών, αλλά και στα αστικά κέντρα να οριστούν συγκεκριμένε ζώνε προστασία για να επιδιώξουμε το σωστό στόχο. Ε, Επίση, επενδύσει στην εκπαίδευση. Καθοριστική σημασία για την καινοτομία, Πρόεδρε, και με αυτό θα κλείσω. Όπω λέει η ισχυώδη μα, τα ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να προωθήσουν την τεχνολογική εκπαίδευση στου νέου και τα παιδιά. Νομίζω αυτό που προσπαθεί να πει είναι ότι η βάση για τη μελλοντική καινοτομία και για την καθαρή ενέργεια είναι οι νέοι. Χρειαζόμαστε λοιπόν δυναμισμό, μια δυναμική προσέγγιση ε, για την καθαρή ενέργεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Θήτο. Ευχαριστώ, και εγώ ε, είναι ευνοϊκά δικείμενο στην γνωμοδότηση της κυρίας Μόλκοβα και θεωρώ ότι όλες τις παρατηρήσεις είναι εύστοχες και αναγκαίες. Συμμερίζομαι τις ανασυχίες της συναδέλφου σε σχέση με την ποικιλομορφία και το περίπλοκο των χρηματοδοτικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται ήδη και πιστεύω ότι σκόπιμο θα ήταν να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να απλωστευτούν και να αλληλοσυμπληρωθούν και να μπορέσουν και οι τοπικές αρχές να έχουν ευκολότερη πρόσβαση στις πηγές χρηματοδότησης. Επίσης συμφωνώ με την ανάγκη βελτίωσης της προσέγγισης της ευφυούς ε, καινοτομίας με καλύτερη χρήση των κονδυλίων και ενίσχυση των σχέσεων συνεργασίας της κοινωτικές πολιτικές, τις εθνικές και τις περιφερικές όλων μεταξύ τους. Τέλο, ε, η γνωμοδότηση σωστά μιλάει για την επιτάχυνση τη μετάβασης σε μια ανταγωνιστικότερη οικονομία που να βασίζεται σε λιγότερη κατανάλωση άνθρακα. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία που πρέπει να την ε, εκμεταλλευτούμε και μπορεί να συνεισφέρει στο να δημιουργηθεί απασχόληση, περισσότερες επενδύσεις και οικονομική ανάπτυξη, καθώς επίσης και να επιδιώξουμε και να πετύχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν το λόγο για τη γνωμοδότηση αυτή. Όχι. Θα δώσω το λόγο στην κυρία, στον κύριο Ντέρλ. από την ε, ερευνητική μονάδα της Κομισάνου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που λάβαμε αυτή την, αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Οι προτάσεις της Επιτροπής Ρέτζη ε, υποστηρίζουν την ε, πρωτοβουλία της Κομισιόν και την ενισχύουν. Και θέλω απλά να αναφερθώ σε ορισμένα σημεία που έχουν ε, τη σημασία τους και που αναφέρθηκαν και στα σχόλιά τους από τα μέλη της Επιτροπής. Όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη, ο κύριος Ντέλη νομίζω είπε κάτι για τις εκπομπές. Ο εξεγνωρισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι πλήρως ενσωματωμένος με βάση τους στόχους ε, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και ε, έτσι οι στόχοι για την καθαρή ενέργεια βεβαίως ε, υπηρετούν ακριβώς αυτούς τους στόχους. Υπάρχουν πολλές αναφορές όσον αφορά τη σημασία του πολίτη και των σχέσεων του πολίτη και πώς μπορεί να ενταχθεί ο ίδιος ο πολίτης σε αυτήν την καινοτομία για την καθαρή ενέργεια είναι βασική μας φιλοδοξία η αύξηση της πρόσβασης και της συμμετοχής των πολιτών, καθώς οι πολίτες είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες για την επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Και ε, γνωρίζουμε ότι ο βαθμός που μπορούμε να επηρεάσουμε τις επιλογές των πολιτών ε, θα επηρεάσει και τον, το βαθμό εκπλήρωσης των στόχων που έχουμε θέσει. Και καθώς βρισκόμαστε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, θα σας πω κάτι που το γνωρίζετε ε, ήδη. Τα σημεία στις παραγράφους 2 και 3 που αναφέρονται σε, αυτά τα, σε, αυτές, δύο παρα, σε αυτές δύο παραγράφους βεβαίως αφορούν τη μετάβαση, ε, την ενεργειακή μετάβαση, ε, την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων κτλ. κτλ. Καθώς αυτό το θέμα έχει σχέση και με τον ανταγωνισμό και με την καλύτερη χρηματοδότηση, η διαχείριση των ε, ταμείων και της χρηματοδότησης θα επέξει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ε, καινοτομία. Όλα αυτά βεβαίως υπηρετούνται και από τις διάφορες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Κομισιόν, αλλά ε, σημαντικές θα είναι οι συμπράξεις που θα ε, δημιουργηθούν ανάμεσα σε διάφορες πλατφόρμες, εξειδικευμένες πλατφόρμες, μεταξύ άλλων και στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Και όλα αυτά ενηφέρονται και στην ανακοίνωση για την, με τίτλο «Ενίσχυση της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο για την ενίσχυση της εδαφικής συνοχής». Επιπρόσθετα προς αυτή την ανακοίνωση υπάρχει ένα ειδικό σημείο το οποίο αναφέρεται ιδίω στις συμπράξεις που αφορά και το, και την, το κέντρο συμβουλευτικής της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, όπου και αναδεικνύεται η ανάγκη να υπάρξει ε, συνδυασμός διαφόρων χρηματοδοτικών πόρων. Πολλοί αναφέρθηκαν στα χρηματοδοτικά μέσα. Και βεβαίω η Κομισιόν γνωρίζει την ανάγκη απλούστευση των χρηματοδοτικών μέσων. Αυτό το ζήτημα ήδη έχει αντιμετωπιστεί σε ένα βαθμό τουλάχιστον στον κανονισμό Omnibus που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο του τριμερούς διαλόγου. Ε, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο βεβαίως θα πρέπει να μας απασχολήσει και στο μέλλον. Τέλο η Κομισιόν ε, συμφωνεί ότι το ευρωπαϊκό θεματολόγιο είναι ο κατάλληλος, ένας κατάλληλος χώρος για την αύξηση της ε, ευαισθητοποίησης και των γνώσεων των πολιτών για αυτό το ζήτημα. Η κυρία Μιλαντίνοβα, ευχαριστώ. Ευχαριστώ την, και τον ε, συνάδελφο από το Κέντρο Έρευνας. Ε, θα προχωρήσω σε κάποιο πολύ συγκεκριμένο τεχνικό σχόλιο. Νομίζω ότι το σχέδιο γνωμοδότησης αντιμετωπίζει πολύ σωστά την, ε, το, το, το, το, ζήτημα της περιφερειακής διάστασης στην πολιτική κυριοτομίας. Απλά στο σημείο 6 για λόγους ε, αποσαφήνισης. Αναφέρεται ότι τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά μέσα και στη συνέχεια τα, τα διάφορα προγράμματα. Ίσως θα μπορούσε λοιπόν να πει κανείς ε, ε, να αναφερθούν μάλλον σε αγγείλες προκειμένου να καταστεί σαφής η διαφορά. Δηλαδή ε, τα, τα, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία και ορίζοντας 2020 είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ίσως θα μπορούσαν κάπως να ξεχωριστούν ε, μέσα στο κείμενο αυτό για να, για να προκύπτει ε, σαφώς αυτή η διάκριση. Ευχαριστώ κύριε Πίκολα. Θέλετε να απαντήσετε ή ε, θέλετε να μας μεταφέρετε σχόλια τη κυρία Μάλκοβα. Όχι. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για αυτή τη συζήτηση και με αυτό περνάμε στο επόμενο σημείο τη σημερινή διάταξη. Ε, έχουμε προχωρήσει αρκετά γρήγορα. Έχουμε λίγο χρόνο λοιπόν. Ε, περιμένουμε ε, περαιτέρω μέλη τη Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη να προσέλθουν εδώ στην αίθουσα προτού προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Εντάξει λοιπόν. Τότε α κάνουμε ένα διαλυματάκι 15 λεπτών προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι θα έχουν όλα τα μέλη της Επιτροπής μας την ευκαιρία να βρίσκονται εδώ στην αίθουσα ε, για τις ψηφοφορίες. Και συνεχίζουμε στις 17 και 25.

στα χέρια μου. Ελπίζω να μην χρησιμεύσει για κακό σκοπό. Λοιπόν, θα, ξεκινήσουμε, θα συνεχίσουμε τώρα με τις ψηφοφορίες. Πρώτο θέμα είναι οι εδαφικές τυπολογίες. Γνωστό και ως τερσέτ. Όπως θα θυμάστε, σκοπός αυτής της πρότασης ήταν η τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού ΝΑΤΣ, προσθέτοντας εδαφικές τοπολογίες που χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως, αλλά αυτή τη στιγμή δεν την χάνουν αναγνώρισης. Αρχικά η Ρέτζη αποφάσισε να ακολούθησει την ε, απλουστευμένη διαδικασία, λαμβάνοντας, υιοθετώντας τη θέση της Κομισιόν χωρίς τροπολογίες. Είχαμε ε, εδώ ε, προσκαλέσει εκπροσώπους της και είχαμε λάβει την ε, απόφαση αυτή. Αυτή ήταν η εντολή που έλαβε η διαπραγματευτική ομάδα στην Ολομέλεια τον Ιούλιο φέτος. Ωστόσο, το Συμβούλιο επιθυμεί να εισαγάγει ορισμένες τεχνικές και όχι αμφιλεγόμενες τροπολογίες. Έγινε λοιπόν ένα τριμερής Διάλογο 26 Σεπτεμβρίου. Εγώ συμμετείχα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, εκπροσωπήθηκε η Εστονική Προεδρία ε, και η Κομισιόν από επικεφαλής μονάδας της Γενικής Διεύθυνσης Eurostat. Με πολύ γρήγορο ρυθμό καταφέραμε να φτάσουμε σε συμφωνία επί ενός κοινού κειμένου στο οποίο θα ενσωματώνονταν οι προτάσεις αλλαγής του Συμβουλίου. Το συμφωνηθέν κείμενο επιβεβαιώθηκε με την συνήθη επιστολή από τον πρόεδρο του Κορεπέρ, την οποία και σας ε, απέστειλα μέσω email και που μπορείτε να βρείτε και στο φάκελό σας σήμερα. Γι' αυτό και ε, θα ήθελα να σας ζητήσω αυτή τη στιγμή να εγκρίνουμε την έκθεση αυτή. Αν εγκριθεί θα προχωρήσει στους ε, νομομαθείς γλωσσολόγους και στη συνέχεια θα ε, διαβιβαστεί στην ε, Ολομέλεια. Λοιπόν, ε, αυτή τη στιγμή αν υπάρχει κάποιος από, εκπρόσωπος του Συμβουλίου, όχι. Από ό,τι φαίνεται, επομένως μπορούμε να προχωρήσουμε στην προφορία επί του συμφωνηθέντου κειμένου που έχετε ήδη λάβει. Μία ψηφοφορία θα γίνει και αυτή θα γίνει ηλεκτρονικά. Παρακαλώ ψηφίστε τώρα. Is The is closed. And Εγκρίνεται. Μπορούμε να προχωρήσουμε όπως περιέγραψα. Το επόμενο θέμα αφορά την έκθεση πρωτοβουλίας της κυρίας Γκαρσία Πέρες ανάπτυξη των μέσων ε, των μηχανισμών πολιτικής συνοχής αναπεριφέρεια για την αντιμετώπιση των δημογραφικών αλλαγών. Έχουμε λάβει 231 τροπολογίες στο σχέδιο έκθεσης αυτό και η συγκήτρια προτείνει κάποιε συμβαστικέ τροπολογίε. Πριν από την ε, ψηφοφορία, πριν προχωρήσουμε στην ψηφοφορία, κυρία Περέζη, θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομη. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ όλους όσοι συνεργάστηκαν ε, στην εκπόνηση και των τροπολογιών αλλά και των συμβαστικών ε, τροπολογιών, τους και εισηγητές δηλαδή, τους συνεργάτες των διαφόρων πολιτικών ομάδων. Όλους τους ευχαριστώ πολύ γιατί με τις προσπάθειές τους βελτιώνεται το κείμενο και παρόλο που εστάλει ένα mail με διορθώσεις για την ψηφοφορία οι αλλαγές η τροπολογία 9 με κατά 36 υπέρ και 185, 86 και 87 ψηφίζω κατά. Είναι πληροφορίες που έχουν οι πολιτικές ομάδες, αλλά ήθελα να το επαναλάβω και να επαναλάβω και τις ευχαριστίες μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα περνάμε στην ψηφοφορία και αρχίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 5. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 54. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Ελέγχουμε για την τροπολογία 54. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Βλέπετε και εσείς τα αποτελέσματα. Τα βλέπετε, τέλεια. Απορρίπτεται λοιπόν. Περνάμε στη συμβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. εγκρίνεται. Τροπολογία 65. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 72. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ας ψηφίσουμε λοιπόν επί της τροπολογίας 73. Παρακαλώ. Ψηφίστε. The vote is closed. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Όχι, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται βεβαίω. Η τροπολογία 73 απορρίφθηκε. Συμβιβαστική τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 89. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Α ψηφίσουμε ηλεκτρονικά λοιπόν επί της τροπολογία 89. Παρακαλώ ψηφίστε τώρα. The vote is closed. Απορρίφθηκε. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ας ελέγξουμε λοιπόν. Θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τώρα επί της τροπολογίας 93. The vote is closed. Εγκρίνεται. Συγγνώμη, ήταν δικό μου το σφάλμα. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 101 υπέρ. 101 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίφθηκε. Θέλετε να το ελέγξουμε, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ας ψηφίσουμε λοιπόν, άρχεται ψηφοφορία τώρα. The vote is It is rejected. Απορρίφθηκε. 102. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. Θέλετε να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ας το ελέγξουμε λοιπόν. Ψηφίστε παρακαλώ τώρα. The vote is closed. The same result. Το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Απορρίφθηκε. Μπορείτε και να το θυμάστε. Να το απομνημονεύσετε. Να το χρησιμοποιήσουμε και σε επόμενες ψηφοφορίες. 105 υπέρ. Κατά αποχές απορρίφθηκε. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 120 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Τροπολογία 146. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 147. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να το ελέγξουμε. Ας το ελέγξουμε. Ας ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά τώρα επί της ε, τροπολογίας 147. Ψηφίστε παρακαλώ. The vote is closed. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. Compromise 15. Συμβαστική 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 157. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ας το ελέγξουμε καλύτερα. Ας ψηφίσουμε λοιπόν επί της τροπολογίας 157 τώρα ηλεκτρονικά. The vote is closed. Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Ήδη ακριβώς αποτέλεσμα. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 164. Υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας το ελέγξουμε καλύτερα όμως με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ας ψηφίσουμε τώρα. Άρχεται ψηφοφορία. The vote is Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συγγνώμη, συγγνώμη. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 176. 176 λοιπόν, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 177 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 18. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 184. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 19. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 191. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 194. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 20. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 21. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 22. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 23. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 24. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 228. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ναι, παρακαλώ. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Την 172, γιατί δεν την ψηφίσαμε. Επαναλαμβάνει στα αγγλικά, μελήτρια. 172. Δεν ξέρω γιατί δεν την ψηφίσαμε αυτή την τροπολογία. The explanation from the Secretariat. Η εξήγηση της Γραμματείας είναι ότι αυτή η τροπολογία καλύπτεται από τη συμβαστική τροπολογία 12. Η συγκεκριμένη. Εντάξει, ευχαριστώ. Και περνάμε στη συμβαστική 1. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Τροπολογία 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ, κατά, αποχές, ας το ελέγξουμε καλύτερα. Ας ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά τώρα επί της τροπολογίας 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is Πέρας Απορρίφθηκε. Με συγχωρείτε πολύ, δικό μου το σφάλμα. Τροπολογία 29. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 40 Θέλετε να ελέγξουμε την τροπολογία 39. Ωραία. Ψηφίστε παρακαλώ επί της τροπολογίας 39 ηλεκτρονικά. The vote is closed. ολοκληρώθηκε και εγκρίνεται. Με συγχωρείτε. Σαράντα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 42 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ, κατά, αποχές, Ας το ελέγξουμε καλύτερα. Ξεκινάει τώρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της τροπολογίας 44. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται να το ελέγξουμε. Ας ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 46 αυτή τη στιγμή. Πέρα. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 47. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας το ελέγξουμε. Ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία αυτή τη στιγμή επί της τροπολογίας 47. Ψηφίστε παρακαλώ. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Με μία ψήφο διαφορά όμως, ε. Μάλλον πρέπει να κάθομαι να μετράω τα χέρια σας, ένα-ένα. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές Ας το ελέγξουμε καλύτερα, μιας και είναι η τελευταία ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά τώρα. The vote is closed. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην ε, τελική ψηφοφορία που θα γίνει ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. The vote is Η έκθεση της Συγχαρητήρια, κυρία Καρσία Πέρες. Thank you. We, we... Συνεχίζουμε τώρα. Και περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία που είναι το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για την περίοδο μετά το 2020. Ο κύριος Βόν είναι ο εισηγητής. Θέλετε να πείτε κάτι? Ναι, σύντομα θέλω να σχολιάσω ε, τη συνεργασία που είχαμε σε σχέση με την έκθεση αυτή. Είχαμε 120 τροπολογίες που καταφέραμε σχεδόν όλες να τις συμπεριλάβουμε σε 13 συμβιβαστικές. Από την ΚΟΕ μέχρι το EFDD. Καταλαβαίνετε ότι χρειάστηκε πάρα πολύ συνεργασία και ε, χαίρομαι που τα καταφέραμε καλά. Ελπίζω περιπομόφωνα να εγκριθεί η έκθεση αυτή, γιατί έτσι θα σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα από την πλευρά μας. Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε για τη συνεργασία όσον αφορά τις συμβαστικές τροπολογίες. Ψηφίζουμε λοιπόν και αρχίζουμε με την τροπολογία ρυθμός τη συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 λέει η πρόεδρος. Α, συγγνώμη, διορθώνει. 4. Συμβαστική 4. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα πάμε στη συμβαστική 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 6. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 8. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πρέπει να ψηφίσουμε τις τροπολογίες 73 και 74, γιατί ζήτησαν χωριστή ψηφοφορία οι πράσινοι. Ωραία. Εμπιστεύομαι τη γραμματεία. Γιατί αυτός είναι ο κανόνας. Ότι δεν μπορούμε να έχουμε χωριστές ψηφοφορίες στις συμβαστικές. Έτσι δεν είναι. Οπότε, αν δεν καλύπτεται και δεν καλύπτεται, τότε μπορούμε να ψηφίσουμε χωριστά. Οπότε ψηφίζουμε τις τροπολογίες 73 και 74 επειδή δεν καλύπτονται από τις συμβαστικές. Τροπολογία 73. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 74. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 11 τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 93. Υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά, τροπολογία 93. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Συμβαστική τροπολογία 12 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 118 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα φτάνουμε στην τελική ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. τέλος της ψηφοφορίας και εγκρίθηκε η γνωμοδότηση. Συγχαρητήρια κύριε Βόχαν. Και σας ε, ευχαριστώ για τη δουλειά σας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Εδώ λίγη η συνεδρίασή μας και συνεχίζουμε με τη συνεδρίαση των συντονιστών. Όσοι δεν συμμετέχουν στη συνεδρίαση των συντονιστών, παρακαλώ να αποχωρήσουν ησύχως.